Άρχεται η Σύνοδο των Εργασιών. Σα καλωσορίζω θερμά όλους στην αίθουσα της Ολομέλειας και θα ήθελα να καλωσορίσω και του εκπροσώπου ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπή που είναι μαζί μα σήμερα και επίση να καλημερίσω όλου του ευρωβουλευτέ που βρίσκονται στην αίθουσα και όλους εκείνου που παρακολουθούν τις συζητήσεις μας μέσω των της τηλεόρασης. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι πολλοί παρακολουθούν από τις οθόνες τους ε, τις συζητήσεις και με πολύ προσοχή. Αλλά και η έμπρακτη συμμετοχή στη συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και σας ε, προσκαλώ θερμά να συμμετέχετε και στις συζητήσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για τις ε, διακοινοβουλευτικές επιτροπές οι ε, προθεσμοί για τις υποψηφιότητες ε, λήγει σήμερα